Συνάδελφοι, επανερχόμεθα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά καθυστέρησε ο Θαλής. Ευχαριστώ τον κύριο Σαβαρμά, ο οποίος με αντικατέστησε και προείδευσε στο πρώτο τμήμα της συνεδρίασης. Επανερχόμεθα λοιπόν και είμαστε όλοι συγκινημένοι ε, συνειδητοποιώντας το δράμα το οποίο χτύπησε την Πορτογαλία αυτές τις μέρες και κατάλαβα ότι ο Φερνάντες θα ήθελε να αναφερθεί στο έβρος του προβλήματος αυτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το Σαββατοκύριακο ζήσαμε μια τραγωδία στην Πορτογαλία. Δυστυχώς ε, Έχουμε 64 επιβεβαιωμένα θύματα, μάλλον δυστυχώς θα υπάρξουν και άλλα. Η πλειοψηφία των θυμάτων αυτών έχασε τη ζωή της ε, από την πυρκαγιά. Έπεσε ένας ε, κεραυνός, ε, χωρίς να ακολουθήσει όμως βροχή και αυτό προκάλεσε μια τέτοια καταστροφή να υπογραμμίσω την ταχύτητα με την οποία ο Επίτροπος Τηλιανίδης και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσαν αυτούς την διάθεση της Πορτογαλίας για να ξεκινήσει τη λειτουργία του ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και για να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί από συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν υπάρξει αίτηση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα κάνει και το Κοινοβούλιο. Αυτό θα είναι μια επίδειξη, αν θέλετε, του αισθήματο της αλληλεγγύης, αλλά και μια υποχρέωση από πλευράς μας μπροστά απέναντι στα θύματα και τις οικογένειες ε, που υποφέρουν και πενθούν. Όλα τα μέτρα λοιπόν τα οποία μπορούμε να πάρουμε σε σεβόμενη ε, μια ευρωπαϊκή πολιτική δασοκομείας η οποία να βασίζεται στην πρόληψη, στην πιθανότητα δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Πολιτικής Προστασίας απέναντι σε ακραία φαινόμενα τα οποία δυστυχώς θα έχουμε μπροστά μας λόγω των κλιματικών αλλαγών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε. Για μια ακόμη φορά λοιπόν αγαπητέ συνάδελφε θα σας πω και νομίζω ότι μεταφέρω τα αισθήματα του συνόλου των συναδέλφων την συμπάθειά μας ε, για αυτό που συνέβη, για τα θύματα και για την χώρα σας συνολικά. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη είναι μια μεγάλη οικογένεια και σε αυτές τις δραματικές στιγμές θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να συνδράμουμε και να ε, δείξουμε με δύναμη και αποφασιστικότητα την αλληλεγγύη την οποία έχουμε. Λοιπόν, επανερχόμεθα θα επανέλθουμε στο σχέδιο κανονισμού το οποίο αναφέρεται ε, στο FC2 και επεκτείνει την προθεσμία την Οι συζητήσεις μέχρι τώρα έγιναν από τις ε, επιτροπές ECON και Budget Μετά από την ψηφοφορία ξεκινάει ένας, μία περίοδος ε, τριγωνικού διαλόγου και ευχαριστώ τον κύριο Σαβαρμά, ο οποίος έχει προεδρεύσει του διαλόγου αυτού και σήμερα θα ακούσουμε τον, Juan Manuel, τον Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες ε, για το πού βρισκόμαστε και τι δυνατότητες έχουμε για να υπάρξει θετική κατάληξη. Ευχαριστώ Πρόεδρε Ευχαριστώ όλους όσους έχουν εμπλακεί στην συζήτηση μέχρι τώρα και την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο που πήραν μέρος ε, στις συζητήσεις αυτές, της τριμερείς, τους εισηγητές, τους σκιώδεις και όλους όσους γενικά πήραν μέρος στην συζήτηση. Εμείς σαν Κοινοβούλιο έχουμε μια ενιαία θέση και σεβόμεθα την εντολή την οποία μας δώσατε. Θυμίζω ότι ο διάλογος αυτός ξεκίνησε στις 31 Μαΐου. Έγινα μια μεικτή συνάντηση, ε, τρεις με έγιναν μέχρι τώρα, θα υπάρξει ένας τέταρτος αύριο. Έχουμε προχωρήσει σε αρκετά σημεία και μπορεί κανείς νομίζω να ελπίζει ότι θα υπάρξει μια νέα τελική εντολή για να καταλήξουμε ε, για την θηρίδα ε, για τις ε, μικρομεσές έχουμε μια δυνατότητα πρόβλεψης εγγύησης η οποία μπορεί να αυξηθεί μετά από την προσθήκη της Διευθυντικής Επιτροπής του Steering Board περιπτώσει και μπορεί να φτάσει τα 9 δις. Αναφέρομαι ε, στην συνεισφορά και τις εγγυήσεις που μπορεί να δώσει ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Οι τομείς τους οποίους καλύπτονται από το ΕΦΣΥ, ε, οι διαδικασίες συμβατοποίησης τους με τις υπόλοιπες ε, διαδικασίες χρηματοδότησης, με τις πλατφόρμες ενημέρωσης και συμβουλών, η τιμολόγηση των δράσεων του ΕΦΣΥ, ο συντονισμός των δράσεων του ΕΦΣΥ, είναι όλα αυτά θέματα τα οποία μπορούν να γίνουν αντικείμενο της τελικής εντολής. Το βαθμολόγιο, οι δείκτες που θα πρέπει να εξετάζονται από την Επιτροπή την Επενδυτική, η αξιολόγηση των επιτευγμάτων, όλα αυτά είναι θέματα στα οποία υπήρξαν κάποια θετικά βήματα αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε τομείς όπως η προσθετικότητα, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις ε, συνθήκες οι οποίες επικρατούν ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, η πρόσβαση στις εγγυήσεις και η δυνατότητα ύπαρξης μιας πιο, ενός πιο δυνατού ρόλου των εθνικών επενδυτικών τραπεζών. Σε όλους τους τομείς αυτούς υπήρξαν βήματα. Υπάρχουν τρία σημεία στα οποία υπάρχουν θέματα. Είναι τρία σημεία. Το πρώτο είναι ε, το θέμα της χρηματοδότησης. Θυμίζω ότι έχουμε 150 εκατομμύρια τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει από τα περιθώρια το Συμβούλιο από πλευράς του στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης ΕΦΣΥ λέει ότι ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει μέσω της ανακατανομής των πιστώσεων. Φυσικά και έχει τεθεί ένα αστερίσκος στη συγκεκριμένη γραμμή, ότι δηλαδή η συμφωνία δεν προκαταλαμβάνει και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς την απόφαση της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής και οι διαπραγματεύσεις οι οποίες τρέχουν δεν έχουν ακόμα καταλήξει, αλλά για τα 500 εκατομμύρια τώρα, τα οποία προτείνει η Επιτροπή να πάρουμε από το Connecting Europe, ε, εδώ για μια ακόμη φορά πρόκειται για ένα σημαντικότατο πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ λέμε μπάστα, ως εδώ και μη παρέκει. Ακόμα και στα πλαίσια του FC1 είχε υπάρξει μια συμφωνία και ήδη είχαν ε, βγει ε, ένα τμήμα των χρημάτων από το Connecting Europe και τότε είχαμε πει και είχαμε συμφωνήσει και πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες ότι δεν θα έπρεπε να αφαιρεθούν περαιτέρω χρήματα από το Connecting Europe. Και όμως δυστυχώς για το FC2 θέλουμε να αφαιρέσουμε από τον προϋπολογισμό του Connecting Europe 500 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει και οι συμφωνίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Πρέπει κανείς να τηρεί τον λόγο του. Και δεν είναι καν αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει υπάρξει μια συμφωνία για το στρατηγικό ταμείο. Εγώ προτείνω λοιπόν να πάρουμε αυτά τα 500 εκατομμύρια από το περιθώριο και εδώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα περάσουμε από 315 ε, ε, δις ευρώ σε 500 δις ε, το ε, στρατηγικό ταμείο έχει κινητοποιήσει 194 δις, έχει βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεων και ε, ακριβώς λόγω αυτών των 500 εκατομμυρίων δεν θέλει να περάσει από τα 3,15 στα 500 δις. Λοιπόν, εφόσον το Συμβούλιο εμένει, θα πρέπει και εμείς να εμείνουμε ε, και δεν θα πρέπει αυτά τα 500 εκατομμύρια τα οποία θα διαιρεθούν για ε, 28 ε, να μην υπάρξει μια τελική επένδυση 500 δις αυτή τη φορά. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της διακυβέρνησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί έναν εκπρόσωπο του στο steering board και οι αποφάσεις ε, θα πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία 4 πέμπτων. Ε, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σε κρεμότητα αλλά έχει υπάρξει κάποια μικρή πρόοδος είναι οι σχέσεις σε φορολογικό επίπεδο με τις λεγόμενες μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες εμείς θα θέλαμε εδώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όχι μόνο να αναλάβει την υποχρέωση να μην έχει σχέσεις ε, με ε, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα, ε, είναι εγκατεστημένες δηλαδή σε μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, αλλά και να ελέγξει τις δικαιοδοσίες στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν. Νομίζω ότι έχει γίνει εδώ κάποια πρόοδος. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να κλείσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Μάλτα. Από πλευράς Κοινοβουλίου κάτι τέτοιο είναι εφικτό και επιθυμητό. Από πλευράς όμως Συμβουλίου και παρά και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό ε, τις προσπάθειες της Προέδρου Δεν είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει μια εντολή για συμφωνία σε μια τέτοια τόσο σημαντική περίπτωση για το Κοινοβούλιο. Από την αρχή το Κοινοβούλιο είναι σαφές, ενωτικό, γνωρίζει τι θέλει, είναι διαθέσιμο για τη διαπραγμάτευση. Όπως είπα η διαπραγμάτευση έχει προχωρήσει και ευχαριστώ την Προεδρία της Μάλτα για όλες τις προσπάθειες τις οποίες έκανε και για τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουν γίνει. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα της χρηματοδότησης όπως και το θέμα της διακυβέρνησης και το θέμα των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, χωρών δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα καταλήξει σε μια καλή συμφωνία. Αν δεν τα καταφέρουμε κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας της Μάλτα, τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε. Νομίζω όμως ότι το Συμβούλιο έχει το ίδιο συμφέρον ε, για επενδύσεις ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι επενδύσεις είναι σημαντικές και για την απασχόληση και για την ανταγωνιστικότητα, όπως επίσης και για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη και τα 28 μεμονωμένα κράτη-μέλη επαναλαμβάνω ήδη, 420.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν στηριχθεί οικονομικά από το Στρατηγικό Ταμείο. Θα πρέπει να βελτιώσουμε, αν θέλετε, την εικόνα που έχει το Ταμείο αυτό, γιατί ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει. Είναι όμως κάτι το οποίο έχουμε βελτιώσει, είναι κάτι το οποίο είναι επιβελτιώσιμο αλλά νομίζω ότι στα σημεία όπου δεν έχει υπάρξει συμφωνία μπορώ να υπολογίζω στην καλή πίστη του Συμβουλίου. Ευχαριστώ τον Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες για τις διευκρινήσεις τις οποίες έκανε. Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις με το Συμβούλιο. Για το θέμα της χρηματοδότησης γνωρίζετε άλλωστε ότι για τη διασφάλιση της κάλυψης των 500 εκατομμυρίων στον τομέα της άμυνας για το 2020 προβλέπεται να πάρουμε πάλι από το Connecting Europe. Οπότε εδώ υποπτεύομαι ότι θα ακολουθήσουν εξαιρετικά δύσκολες συζητήσεις. Ποιος θα ήθελε το λόγο, η Αίντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Γιατί στηρίζουμε απολύτως τη θέση του Ζωζέ Μανουέλ. Και ο Ούντο Μπούλμαν τα ίδια είπε εκπροσωπώντας εκεί το κοινοβούλιο με σαφέστατη εντολή ε, για τις διαπραγματεύσεις και πολύ μεγάλη υποστήριξη των δύο επιτροπών του κοινοβουλίου. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό διαπραγματεύονται. Τα περισσότερα θέματα από πρότεινε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διευκολύνει κατά τα άλλα πολύ τη δουλειά, πάντα κάνει προτάσεις επικοδομητικές, συμβιβαστικές, και υιοθετεί πολλές φορές ε, πολλές από τις θέσεις μας. Αλλά για άλλη μια φορά στο θέμα της χρηματοδότησης προσκρούμε σε τείχο το Συμβούλιο. Από ό,τι φαίνεται επιτέλους θα αρθεί το βέτο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου. Ελπίζω αυτό να δώσει μια νέα πνοή φρέσκια έτσι, στο Συμβούλιο και να τους φωτίσει ε, να δούνε διαφορετικά τις διαπραγματεύσεις. Βεβαίω, τα 500 δι είναι λεφτά πολλά, όπως λέει και ο Σωσέ αν αρχίσουμε να τα διαιρούμε με τι χώρε και τα χρόνια δεν είναι και τόσα πολλά. Και αν έχει τέτοια επιτυχία το σχέδιο Juncker, το επενδυτικό που έχει και γι' αυτό το στηρίζουμε και είναι για φόρου και θέλουμε και να παραταθεί ε, και να διευρυνθεί, θα πρέπει να κάνουν και μια προσπάθεια τα κρατη Το ίδιο με το Connect Europe Facility. Τι γίνεται για αυτή, με αυτή τη διευκόλυνση. Τι έγινε αυτό το πρόγραμμα, το εφήβραμε για να πηγαίνουμε να παίρνουμε για τα υπόλοιπα στο FC1, στο FC2, στην άμυνα. Περάστε κόσμο. Και δεν έχει και το Connect Europe ε, μεγάλη πρικοδότηση για το ύψος των υποδομών που χρειάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. βγάζουμε λεφτά από τη μία τσέπη για να τα βάλουμε στην άλλη. Ελπίζω στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου να ε, δώσουμε λίγο περισσότερο οξυγόνο σε όλη αυτή την υπόθεση. Άλλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Χωσέ Μανουέλ μας έδωσε μια πολύ καλή επισκόπηση της κατάστασης. Δεν έχω λοιπόν πολλά να προσθέσω, αλλά θα ήθελα να τονίσω το εξή. Όταν ξεκινήσαμε με το πρώτο έτσι, καταλάβαμε τη στρατηγική του σημασία. Και γι' αυτό Ήδη στον πρώτο γύρο προσφέραμε, χρήματα, προσφέραμε πόρους από τον προπολογισμό. Η ηρωνία τώρα είναι ότι όλοι λένε ότι είναι εξαιρετικά καλό το πρόγραμμα αυτό, αλλά τα κράτη-μέλη αρνούνται να συνεισφέρουν. Και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πόσο στενοκέφαλη μπορεί να είναι. Εάν δεν ενδώσουν, ας το κλείσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος το Συμβούλιο μόλις δέχτηκε την αναθεώρηση. Ενημερωτικά μαθαίνω ότι δέχτηκε την αναθεώρηση το Συμβούλιο. Άρα θα πρέπει να απευθύνουμε ένα φόρο τιμής στη Βρετανική κυβέρνηση που μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Όχι μόνο για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τον Brexit, αλλά για να συμφωνήσει επίσης για την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ. Δεν, είναι μόνο Βρετανοί. Ε, ε, νομίζω ότι η, η, δεν ήταν ομόφωνη απόφαση, αλλά οι Ιταλοί και οι Βρετανοί ε, απήχαν. Καλά, η σιωπή του εκλαμβάνεται ω συνένεση. Πριν δώσω το λόγο στον Ζωζέ Μανουέλ για τις μη συνεργαζόμενες ή συνεργάσιμες δικαιοδοσίες. Δηλαδή αυτό είναι η φορολογική παράδειση. Οι μαύρες τρύπε της φορολογίας. Εκεί θα πρέπει να είμαστε απόλυτα κατηγορηματική. Και το Συμβούλιο και η Προεδρία Μαλτέζικη θα πρέπει να είναι αποφασισμένη να τα πολεμήσει. Εγώ δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Οτιδήποτε ε, συνιστά ε, καταχρηστική βελτιστοποίηση και φοροαποφυγή θα πρέπει να πατάσετε και να είμαστε απόλυτοι και δημόσια και στην Ολομέλεια. Αυτό ενδιαφέρει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Ζωζή Μανουέλ. Συμφωνώ απόλυτο. Ελπίζω να σας ακούει και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Όπως είπα και προηγουμένως είναι πάρα πολύ ενωμένο το Κοινοβούλιο και ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία με τον άλλο συνεισηγητή, τον Ούντο Μπούλμαν. Επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσω για την πάρα πολύ επικοδομητική στάση ε, πιστή και παραγωγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προσπαθεί να βοηθήσει την κατάσταση και πραγματικά βοηθάει. Με καλές προτάσεις, με επικοδομητικό πνεύμα, με καλές συμβαστικές ε, λύσεις και όπως πάντα το Συμβούλιο δεν δείχνει την ίδια στάση. Τέλος. Ωραία. Ας ελπίσουμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το τριμερή διάλογο χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Βεβαίως, όλα αυτά, στο F1 υπάρχει ένα περιθώριο δανειοδότησης, αλλά δεν θα πρέπει να αργήσουμε να εγκρίνουμε το δεύτερο F. Τώρα θα περάσουμε στην νότια όχθη της Μεσογείου, να δούμε τι έγινε στη Μεσόγειο, θα μας, στην Τυνησία, Θα μας τα πει η Αίτερ που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας σε αποστολή εκεί 21 με 25 Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω αυτές τις τρεις μέρες και κάτι που ήμασταν στη Τινησία. Πάρα πολύ εντατική αποστολή, όπως συνήθως οι αντιπροσωπείες από τις 7 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Χωρίς λεπτό, ούτε ανάσα δεν πέραμε. Έτσι γίνονται οι αποστολέ και αυτό και είναι ο στόχο, να μην χάνουμε χρόνο και να εκμεταλλευόμαστε και να αξιοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο τις μέρες που είμαστε εκεί για να έχουμε επαφέ, συναντήσει με τι κυβερνήσει, τι ε, οργανώσει, και να βλέπουμε τα έργα που χρηματοδοτεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός Ιδής Όμαση. Έξι βουλευτές πήγαμε εκεί και προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στα έργα αυτά ακριβώς που χρηματοδοτήθηκαν από το μέσο της γειτονίας και αυτά που έχουν να κάνουν με τη διευκόλυνση της γειτονίας. Δηλαδή το έμβριο αυτού που θα αποτελέσει το επόμενο επενδυτικό πρόγραμμα για τις εξωτερικές επενδύσεις. Για να καταλάβετε λίγο το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί από το 2011 μέχρι το 2016 με επιδοτήσεις ε, της τάξεως 1,2 δις και μέχρι το 2020 αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και ο πολιτικός διάλογος που γίνεται, θα δοθούν και άλλα ποσά και μάλιστα θα αυξηθεί κατά 300 εκατομμύρια ετησίω η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 11 μέχρι το 16 δώσαμε 800 εκατομμύρια σε μακροοικονομική βοήθεια, άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σημαντικό εταίρος, σημαντικότατος για τους τινήσιους. Είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εφόρων και Βιώσιμων Επενδύσεων και ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ γιατί ήταν η Τινησία θα μπορούσε να ε, εποφεληθεί από τις επενδύσεις αυτές και ε, τους ενδιάφερε πάρα πολύ η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, περιβαλλοντική πολιτική, όλα αυτά, ε, οι επενδύσεις στις ΑΠΕΣ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί η χώρα έχει μεγάλο δυναμικό και χρειάζεται επενδύσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της επίσκεψης ή της αποστολής εκεί, προφανώς μας συνόδευαν μέλη της αντιπροσωπείας εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας έκαναν ένα πρώτο briefing, μια ενημέρωση πληρέστατη όταν φτάσαμε και ο πρέσβης ε, και ο αντιπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει πάρα πολύ ε, καλή δουλειά. Ξέρουν πολύ καλά τα πράγματα και έχουν μεγάλη παρουσία είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των ε, χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων, ΜΚΟ και τα λοιπά, ε, της κοινωνίας των πολιτών και μάλιστα όχι μόνο οι άνθρωποι της αντιπροσωπείας, αλλά και τα ίδια τα γραφεία είναι ένας κόμβος, είναι σημείο συνάντησης όλων αυτών των οργανώσεων, φορέων, ενδιαφερομένων, δικαιούχων κλπ. Επιχειρήσεις ό,τι και να είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ δραστήρια η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί και ε, προετοίμασαν πολύ καλά την αποστολή μαζί με τη δική μας γραμματεία με τρόπο πάρα πολύ ε, καλό και πληρέστατο. Δέκα συνεδριάσεις είχαμε περίπου. Είδαμε από τον πρόεδρο της Βουλής, μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, επίσης βουλευτές της Ειδικής Επιτροπής Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χρηστής Διακυβέρνησης Καταπολέμησης Διαφθοράς και έλεγχου, ελέγχου της Δημόσιας Δαπάνης. Όλα αυτά είναι μια επιτροπή και είναι πολύ σημαντική για εκείνους. Συναντηθήκαμε και με τον Υπουργό Ανάπτυξη Διεθνούς Συνεργασίας Επενδύσεων και εδώ και λίγες μέρες έχει αναλάβει και Υπουργό Οικονομικών γιατί έγινε ανασχηματισμός. Επίσης, συναντήσαμε το γραφείο του Υπουργού ε, Τοπικών και Περιβαλλοντικών Υποθέσεων. Τώρα προετοιμάζουν τις δημοτικές εκλογές και όλη την αποκέντρωση στην Τινησία. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να ε, συνεδριάσουμε με το Κουαρτέτο Εθνικού Διαλόγου, που ξέρετε ότι είναι τέσσερις εκπρόσωποι τεσσάρων ε, φορέων, εργοδοσία, εργαζόμενοι, τώρα να δούμε θα τους θυμηθώ και τους τέσσερις, αυτοί που πήραν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2015, εν πάση περιπτώσει. Και επίσης ε, είδαμε και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και μας εντυπωσίασε πάρα πολύ η συζήτηση που είχαμε μαζί τους, γιατί είναι πάρα πολύ δραστήριοι θέλουν να ελέγξουν με την κυβέρνηση, αλλά να βοηθήσουν για να πετύχει αυτή η μετάβαση ε, με το σωστό τρόπο στο σωστό δρόμο. Επίση και με διεθνεί οργανισμού συναντηθήκαμε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ΜΠΕΡΤ, η Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη κτλ. Αυτέ ήταν οι συνεδριάσει. Μετά επισκεφθήκαμε και πάρα πολλά έργα. Από ένα κέντρο κράτηση, α πούμε, το οποίο ε, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξυγχρονίζεται εμείς δεν στηρίζουμε απλώς οικονομικά, αλλά βοηθάμε τη χώρα στη διαδικασία της μετάβασης του πολιτεύματος. Δηλαδή αλλάζει και όλη η σοφρονιστική πολιτική και ε, τα δικαιώματα των κρατουμένων, η φροντίδα που παρέχει τους κρατουμένους. Δεν είναι μόνο το κτίριο που ανακαινίζεται εκεί ε, στη φυλακή. Θα πρέπει να ε, ανταποκρίνεται σε κάποια ελάχιστα διεθνή κριτήρια. Λοιπόν, εκεί είναι σημαντική η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήγαμε σε μια αυτοκίνητο βιομηχανία ε, που είναι χειροποίητα αυτοκίνητα ουσιαστικά. Ε, είδαμε κάποιες συνοικίες ε, που ήταν ουσιαστικά παραγκουπόλεις και τώρα υδροδοτούνται, ηλεκτροδοτούνται και έχουν και αποχέτευση. Πήγαμε σε μια επιχείρηση μικροδανείων, μικροπιστώσεων και είδαμε και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν, δύο γυμνάσια, ε, τα οποία επίσης εξεχρονίζονται με το blending, δηλαδή ένα τμήμα των χρημάτων ήταν επιδοτήσεις και ένα τμήμα από την ε, KFW και το Ταμείο Επενδύσεων και στο ΣΦΑΞ που είναι γνωστή μεγάλη πόλη στη Μεσόγειο, η Λιμάνη, είδαμε μια περιοχή που ήταν ε, πάρα πολύ μολυσμένη, δεν μπορούσε κανείς να πατήσει και προχώρησαν στην, στον καθαρισμό από ρήπανση ουσιαστικά για να δούμε πώς αναπτύσσεται όλη η περιφέρεια. Επίσης, είδαμε και σε ένα χώρο co-working, δηλαδή που έχει βραβευτεί, δεν θυμάμαι το Time, κάποιο περιοδικό τους έχει βραβεύσει το People, ότι είναι ο τρίτος καλύτερος χώρος παγκοσμίως ε, εργασίας σε co-working. Τη μέρα που φτάσαμε ή την επομένη, δεν θυμάμαι, τη Δευτέρα, το σκάφος Σαν Τζούστο ε, είχε ε, δέσει ε, στο λιμάνι της Τινιδάς. Ε, έχει ευρωπαϊκή σημαία, καλά ιταλική, αλλά είδαμε το πλήρωμα. Συμμετέχει στην αποστολή Σόφια ε, μας είπαν ότι ε, κάνουν περιπολίες στις λιβικές ε, ακτές για να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο όπλων και τη διακίνηση ανθρώπων. Και μιλήσαμε και με έναν Πορτογάλο ναυτικό, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν σε αυτό το σκάφος, αλλά γενικά υπηρετεί σε υποβρύχιο που κάνουν και αυτά περιπολίες στις λιβικές ακτές. Ε, αυτά, έτσι, για να καταλάβετε ότι είχε από όλα το πρόγραμμα στις τρεις μέρες. Ήταν πολύ θετική η εντύπωση που αποκομίσαμε. Η χώρα ε, είναι τρία χρόνια σε μετάβαση και μετασχηματισμό, παρόλο που απομένουν πάρα πολλά να γίνουν, είναι γεγονός ότι έχουν κάνει μεγάλες πρόοδους για τη σταθεροποίηση και τον εκδημοκρατισμό προετοιμάζουν τις ε, τοπικές εκλογές είναι ε, εντυπωσιακή η συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις, στην εργασία και η διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών. Οι επιπλέον θεωρούν ότι η συμμετοχή αυτή μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα στη χώρα, άρα στηρίζουν ε, τις γυναίκες. Επίσης, ξέρουν ότι πρέπει οι νέοι να συμμετέχουν περισσότερο. Όπως είπαμε, η κοινωνία των πολιτών είναι πάρα πολύ ε, δραστήρια και στον έλεγχο της κυβέρνησης αλλά και στη στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Και είδαμε και κάποια αγωνία μεταξύ των νέων κυρίως, γιατί θέλαν οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις να γίνουν πιο γρήγορα. Και έχουν αρχίσει να αμφιβάλλουν, άξιζε τον κόπο αυτή η επανάσταση. Έπιασε τόπο, θα βγει τίποτα από όλα αυτά, γιατί είναι τεράστια η οικονομική κρίση μετά τις, ε, τα τρομοκρατικά χτυπήματα έχει πέσει κατακόρυφα ο τουρισμός που είναι σημαντική πηγή πλούτου για τη χώρα. Και η οικονομική διακυβέρνηση είναι αρκετά συζητήσιμη της κυβέρνησης, τεράστιο το έλλειμμα, δεν πάει καλά η οικονομία, οπότε οι νέοι κυρίως ανησυχούν και σου λένε εμείς κάναμε την επανάσταση βεβαίως για την ελευθερία αλλά θέλουμε να έχουμε και ένα μέλλον στη χώρα μας. Και εκεί ε, κάπως ταλαντεύονται και αυτή η αστάθεια και η αμφιβολία είναι λίγο επικίνδυνη. Εμεί κατανοούμε αυτέ τι αγωνίε του, το είπαμε, αλλά είπαμε ότι θέλει και υπομονή. Δεν μπορεί να διακυβευτεί όλη αυτή η διαδικασία εκδημοκρατισμού μέσα σε τρία χρόνια. Τρία χρόνια πολύ μικρό διάστημα. Και έχουν γίνει πρόοδοι πάρα πολύ σημαντικέ. Άλλο. Πού είδαμε. Ε, έχει αναλάβει δράση η κυβέρνηση στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Μπορεί να ήταν η λαϊκή κατακραυγή, υπάρχει μεγάλη διαφθορά και ενεργητική και παθητική, γνωστή ήτανε και πέσαν και κάποια χοντρά κεφάλια ε, από δίκτυα και συνδέσεις έτσι, και ο κόσμος ε, αυτά τα χειροκρότησε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πάρα πολύ. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικότατη παρουσία και σημαντικότατο έργο. Διάλογο ε, για βοήθεια και πολιτική χρηματοδότηση έργων. Είναι απίστευτο ο τρόπο με τον οποίο η Τινησία, η Τινήση και η κυβέρνηση έχουν στραμμένο το βλέμμα του προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά δεν ζητούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω γεωγραφική θέση δεν μπορούν, αλλά αισθάνονται σχεδόν Ευρωπαίοι και θέλουν να συμμετέχουν σε όλα. Γιατί θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πλαίσιο σταθερότητα, βοήθεια και δημοκρατικών εγγυήσεων και πολιτική βελτίωση. Και θέλουν να συνεχίσουμε να τους βοηθάμε. Κάτι άλλο που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και τελειώνω η Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιπροσωπεία και έχει σαφέστατη στρατηγική για το τι χρειάζεται να γίνει, όχι μόνο για τις επενδύσεις, αλλά και αυτή η πλαισίωση βοήθεια για τις μεταρρυθμίσεις. Τέλειωσα. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η αποστολή, πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από πρώτο χέρι και να ε, διαπιστώσουμε και να τσεκάρουμε ότι αυτά που κάνουμε εμείς εδώ τα βλέπουν εκείνοι με μεγάλο δεσοσκόριο φαλμού και τα συμμερίζονται και τα εφαρμόζουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την ε, ενημέρωση και για τις θετικές απόψεις τις οποίες εκφράσατε στα πλαίσια της συνεργασίας. Είχατε συνοδευτεί από τον Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες και από την κυρία Βάιντερ. Δεν ξέρω αν έχουν κάτι να προσθέσουν. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Μεταφέρατε αυτά τα οποία συνέβησαν με τον πιο πιστό τρόπο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, όχι. Ε, για τον τουρισμό έχει ανακάμψει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Από ό,τι φαίνεται ότι υπήρξε μια αύξηση κατά 40% το 2016 και προβλέπεται ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και φέτος. Υπάρχει ανησυχία όμως γιατί στο νότο της χώρας αυτή την εβδομάδα υπήρξαν ορισμένες ταραχές και αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να σκιάσει λίγο τα του τουρισμού και μια οικονομία η οποία εξαρτάται τόσο πολύ από τον τουρισμό δεν μπορεί να, α, υποστεί για μια ακόμη φορά. Εμείς στην επίσκεψή μας δεν είχαμε κανένα αίσθημα ανασφάλειας, είναι μια χώρα φιλόξενη και ήμασταν απόλυτος ελεύθεροι. Η κυρία Κρέσλε, σας ευχαριστώ πολύ για την αναφορά αυτή. Συμμετείχα κατά την προηγούμενη αποστολή της Επιτροπής ε, προϋπολογισμού στην Τινησία και θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με την Ισλαμοποίηση. Εμάς μας έκανε εντύπωση αυτό πριν κάποια χρόνια και ε, αρκετές μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, είχαν παραπονεθεί γι' αυτό, διότι ήταν κάτι νέο για την Τινησία. Μπορείτε να μας πείτε πώς το εκτιμάτε, βλέπετε να αυξάνεται ή να μειώνεται. vous s'il vous plaît. απαντήσετε, η κυρία Βάιντερε. Έχετε ζητήσει το λόγο. Ναι, ήθελα απλά να πω λίγα λόγια. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καρδιά Θαπάλε για τον πολύ ικανό τρόπο με τον οποίο ηγήθηκε της αποστολής μας. Τα βασικά ήδη υπόθηκαν. Μου έκανε πολύ εντύπωση, δεδομένου το ότι πρόκειται για πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, ο τρόπος που αντιμετωπίζει το θέμα ε, των αποβλήτων. Επισκεφτήκαμε μια περιοχή τουριστική που ήταν όλα καθαρά, αλλά Λίγο πιο πέρα υπήρχαν βουνά από απορρίμματα ε, στους δρόμους, ε, στις παραλίες παντού. Αυτό είναι απαράδεκτο. Φαίνεται κρίμα να χρηματοδοτούμε ε, τα πανηρά έργα δίπλα, ενώ οι Τινήσοι δεν κάνουν σωστή διαχείριση των απορριμμάτων τους. Και ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε την, ε, την Ισία πιο ελκυστική για τους τουρίστες είναι να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Εγώ, αν ήμουν τουρίστρια, δεν θα ήθελα να πάω εκεί, διότι δεν θα μπορούσα να απολαύσω την ομορφιά της φύσης αν ε, υπάρχουν σκουπίδια παντού. Όπως είπε και η Αίτερ, είχαμε γενικά θετική εντύπωση η επιχειρηματικότητα αυξάνεται με τη δική μας ε, βοήθεια. Νομίζω ότι κάνουμε καλή δουλειά στο θέμα αυτό. Και προσωπικά δεν είδα υπερβολικά επίπεδα Ισλαμοποίησης. Ευχαριστώ. Πριν ε, δώσω το λόγο, Ιντερ, για να δευτερολογήσετε και να κλείσετε, Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Φρανσέσκα Τζίλη, που εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Γειτονία και η κυρία Κριστίνα Φερμέρ, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, θα ήθελαν κάτι να πούν. Έχετε να συμπληρώσετε τίποτα, καμιά παρατήρηση. Ποια κυρία θέλει να λάβει το λόγο, κυρία Τζίλη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να το συνδέσω αυτό με την συζήτηση στην Επιτροπή Κοντ την επόμενη εβδομάδα, όπου θα τεθεί το θέμα του ελεγκτικού συνεδρίου για τη χρηματοδότηση της Τινησίας. Σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή είναι θετική και επιβεβαιεί τις απόψεις τις οποίες εξέφρασαν τα μέλη της, της δικής σας Επιτροπής. Απλά θα ήθελα να συνδέσω αυτά, τις δύο, αυτές τις δύο επιτροπές και τις ευθύνες τους, τις αρμοδιότητές τους. Είμαι, λέγομαι Φαμέιν, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Par les collègues du Parlement qui, qui ont visité la Tunisie. Donc c'est vraiment un sujet prioritaire. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι κατά προτεραιότητα θέματα στις σχέσεις μας με την Τινησία. Στην ανακοίνωση λοιπόν η οποία έγινε από την ύπατη εκπρόσωπο της 29ης Σεπτεμβρίου θα τεθούν τα θεμέλια για την πολυετή βάση της συνεργασίας μας στο μέλλον με την χώρα αυτή για την υποστήριξη των νέων. Ευχαριστώ. Η Άιντερ για να κλείσει η συζήτηση. Να απαντήσω στην κυρία Γκρέσλα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει μια σύγκριση ανάμεσα σε αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα και σε αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν, αλλά σε επίπεδο πέραν του δημοσιονομικού δεν τέθηκαν διάφορα προβλήματα, δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Εμείς συζητήσαμε τα προγράμματα, συζητήσαμε και με εκπροσώπους των Ισλαμικών κομμάτων ή και των μη θρησκευτικών κομμάτων δεν είδαμε εμείς στοιχεία ισλαμοποίησης της δημόσιας ζωής. Υπάρχουν βέβαια κάποια ριζοσπαστικά κινήματα τα οποία είναι ισχυρά κυρίως στο νότο της χώρας. Ήταν ένα κανονικό ταξίδι χωρίς ιδιαίτερες ε, δυσκολίες. είναι μια χώρα Ισλαμική στην πλειοψηφία της, αλλά δεν αισθανθήκαμε εμείς ότι υπάρχει μια προϊούσα Ισλαμοποίηση, μια αλλαγή ως προς το τομέα αυτό. Αλλά αυτός δεν ήταν ακριβώς ο στόχος αυτής της αποστολής, δεν ήταν το βασικό μας θέμα. Δεν ξέρω αν ο Ζωζέ Μανουέλ ή οι Ινές έχουν μια διαφορετική αντίληψη γι' αυτό. Ζωζέ Μανουέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω απολύτως ε, με την Άιντερ. Η Τινησία είναι ένα σημαντικότατος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην το ξεχνάμε. Ε, είναι επίσης η Τινησία ένας σύμμαχος και η επιτυχία αυτής της νέας δημοκρατίας στην χώρα αυτή είναι ουσιαστική για μας. Είναι κάτι που δείχνει ότι στον μουσουλμανικό κόσμο μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία. Υπάρχει η δημοκρατία. Είναι κάτι το εφικτό και υπαρκτό. Υπάρχει επίσης το θέμα της γυναίκας στην κοινωνία αυτή και στην πολιτική γενικότερα Λοιπόν, στο Κοινοβούλιο το 40% είναι γυναίκες. Στις εκλογές οι οποίες θα οργανωθούν για τις τοπικές αρχές, το 50% επαναλαμβάνω θα είναι γυναίκες, είναι υποχρεωτικό και θα υπάρχει ακριβώς το ίδιο ποσοστό σύντομα και στην εκτελεστική εξουσία. Όταν έχετε ας πούμε ε, πρόεδρο άνδρας ε, στην Εθνοσυνέλευση ε, θα πρέπει να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν ένα πραγματικό άνοιγμα, ένας πραγματικός εξυγχρονισμός και επίσης υπάρχουν και υποχρεωτικά ποσοστά εκπροσώπησης των νέων στους εκλογικούς καταλόγους. Η Τινησία έχει βέβαια προβλήματα και κάποια από τα προβλήματα αυτά πρέπει να βρουν σύντομα λύση αλλά βρίσκεται στον σωστό δρόμο και θα πρέπει να υπολογίζει στην δική μας υποστήριξη αλληλεγγύη. Ελπίζω ε, τελικά η Τινησία να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα και για άλλες χώρες έτσι ώστε να δούμε ότι η δημοκρατία και ο Ισλαμικός κόσμος μπορούν να συνυπάρξουν. Το θέμα είναι το ποιος θα προασπίσει την αξία της ανθρώπινης φύσης περισσότερο. Κοιτάξτε όλοι γνωρίζουν ότι ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη στην Τινησία. Καλώς αυτά κλείσαμε με το θέμα αυτό. Θα παρουσιάσουμε τώρα στην έκθεση Βάνα για το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για την περίπτωση της η λεων Κυρία Βάνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, η Ισπανία έχει κάνει αίτηση ε, για ε, συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση στον τομέα εξόριξης του λιχνίτη στην περιφέρεια Καστήλια ή Πέντε επιχειρήσεις αφορά το αίτημα και θα γνωρίζετε ότι στον κανονισμό προβλέπεται να είναι τουλάχιστον 500 οι απολύσεις. Η Ισπανία όμως αιτιολογεί επαρκώς το ε, το ότι έχει λιγότερους ε, απολύσεις λέει ότι ε, οι απολυμμένοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές και γι' αυτό μπορεί να θεωρηθεί η περιοχή αυτή πιο περιορισμένη αγορά. Η Ισπανία ε, ζητάει υπηρεσίες για μέχρι 125 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. οι οποίοι ε, κατά την υποβολή της αίτησης ήταν κάτω των 30 ετών. Υπολογίζει λοιπόν ε, γύρω στα 464 άτομα συνολικά. Η Ισπανία αιτιολογεί το αίτημά της ως εξής. Θεωρεί ότι η ότι ο ευρωπαϊκός τομέας ε, εξόριξης ε, έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις ε, εισαγωγές από τρίτες χώρες. Από το 2005 μέχρι το 2010 μειώθηκαν η ζήτηση στην Ευρώπη λόγω των μεγάλων εξαγωγών από τρίτες χώρες. Και η μείωση αυτή στην Ισπανία ήταν ιδιαίτερα έντονη. Και μάλιστα ε, η συγκεκριμένη περιοχή επηρεάστηκε κατά 80, με μείωση 86%. Ε, έχουν ε, ζητηθεί συνολικά ε, ένα εκατομμύριο 2.264 ευρώ, ε, κάτι παραπάνω δηλαδή από ένα εκατομμύριο ευρώ. Προβλέπεται λοιπόν ε, εκπαίδευση και η στήριξη κατά την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Πολύ θετικό στην επιστολή της ΕΜΠΛ είναι κατά τη γνώμη μου ότι στα μέτρα που προτείνονται προβλέπεται και κάλυψη για την φροντίδα των συγγενών ώστε αυτοί που ε, φροντίζουν ε, άλλα άτομα να μπορέσουν να συμμετάσχουν ε, στο πρόγραμμα αυτό. Ε, τα είναι οι γυναίκες εδώ πέρα και η υποστήριξη των 125 νέων όμως ε, δημιουργεί τη δυνατότητα να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι Φυσικά καλούμε την Ισπανική κυβέρνηση κατά την εφαρμογή των μέτρων να λάβει υπόψη την Συμφωνία του Παρισιού. δηλαδή ε, να στηριχθούν ε, οι προσπάθειες ε, ώστε να καταρτιστούν οι άνθρωποι αυτοί σε βιώσιμες θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι τέτοιες θέσεις εργασίας θα είναι και πιο ανθεκτικές όσον αφορά την μεταφορά σε χώρες χαμηλότερων αμοιβών. Άλλωστε και ε, η οικολογική ε, αυτή η κατεύθυνση αποτελεί στόχο και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Επίση. Σα ευχαριστώ πολύ. Γιατί... Και παρακαλώ να συμφωνήσετε με την έκθεση. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις έχετε, σχόλια έχετε. Όχι. Τροπολογίες για την έκθεση της κυρίας Βάνα. Ποιο ζήτησε το λόγο. Α, ο κύριος Πενίτου Σουλουάγκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση την κυρία Μόνη Καβάνα. Εμείς θα υποστηρίξουμε την ε, ενίσχυση αυτής της περιοχής που έχει πληγεί τόσο σφοδρά από την κρίση. Βεβαίως θα πρέπει να ποντάρουμε σε ένα διαφορετικό, ριζικά ε, διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Εκεί είναι μονοκαλλιέργεια, ε, είναι αποκλειστική η δραστηριότητα τα ανθρακοριχεία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, να σταματήσουμε να και άνθρακα ε, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, θέλω να πω μόνο δύο λόγια ε, και θα κάνω τροπολογίες. Γιατί αυτά μας τα έχουν πει τα συνδικάτα της περιοχής εκεί. Πρώτον, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μια μελέτη για τη ζήτηση εργασίας. Ποιοι είναι οι οικονομικοί τομείς και οι παραγωγικοί τομείς που ενδείκνυνται ε, για να υπάρξει ένα στοιχειώδης επαγγελματικό προσανατολισμός για να στραφούν οι νέοι προς τις κατευθύνσεις αυτές. Και δεύτερο που ζητούν τα συνδικάτα να υπάρχει έλεγχος στη διαχείριση αυτών των ε, ταμείων, να συμμετέχουν δηλαδή και πολίτες ε, και πρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών στη διαχείριση. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Στέφαν Εκ. Ο Στέφαν Εκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κατάσταση είναι πολύ ε, σοβαρή γιατί τα τελευταία έξι χρόνια έχουν κλείσει δέκα εξορεκτικές εταιρείες παρά το γεγονός ε, ότι δεν ανταποκρίνεται απολύτως στον αριθμό των 500 απολυμμένων ε, η συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ την υποστηρίζω γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη και είναι η τρίτη αίτηση κατά σειράν που υποβάλλουν ε, από πλευρά της Ισπανικής Κυβέρνησης το 2017 και μόνο. Θα ήθελα επίσης να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονό ότι οι προτινόμενες δράσεις θα υποστηριχθούν και από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Δηλαδή η αίτηση αυτή δεν είναι μία ε, για την περιφέρεια αυτή. Υπάρχει και άλλη υποστήριξη. Λοιπόν, λαμβανωμένη υπόψη όλων των ε, περιστατικών και των καταστάσεων, υποστηρίζω το αίτημα αυτό. Κυρία Βάνα, έχετε να προσθέσετε τίποτα, καμία παρατήρηση, όχι. Ωραία. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Λίγη ε, σήμερα στις 6 ώρα. Στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε στις 29 του μηνός εδώ στον προπολογισμό και στην Ολομέλεια κανονικά στη Σύνοδο του Ιουλίου. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γιένς Γκάιερ για να μας ενημερώσει για τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλάμε για, ε, τον, ε, για τη συνεργασία των ε, ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και αναδιατύπωση του σχετικού κανονισμού που είναι απαραίτητη. Ε, σύμφωνα με την δέσμη μέτρων ε, καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους. Επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Ήτρε. Το θέμα είναι πώς μπορεί να λειτουργήσει ομαλά η ε, εσωτερική αγορά ενέργειας και πώς μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ε, ε, του μέλλοντος. Σημασία λοιπόν για όλα αυτά έχει ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και αυτό λαμβάνεται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την αναδιατύπωση. Στην Επιτροπή μας ε, κυρίως ασχολούμαστε με τα θέματα διαχείρισης ε, και την οικονομική πλευρά. Ο Έισερ, ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών, ε, θα έχει επιπλέον καθήκοντα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθέσει στο μέλλον, θα πρέπει να μπορεί στο μέλλον να αναθέτει επιπλέον αρμοδιότητες στον οργανισμό αυτόν. Όσον αφορά το, τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, προβλέπεται αυξημένη συνεργασία των διαχειριστών των δικτύων. Αυτό είναι κυρίως το αντικείμενο που θα πρέπει να ρυθμίζει ο Acer στο μέλλον. θα είναι κατά κάποιο τρόπο κόμβος. Και ο Acer θα πρέπει να έχει τους απαραίτητους πόρους ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του. Στο πλαίσιο αυτό, Υποβάλλω κάποιες προτάσεις ε, στο σχέδιο γνωμοδότησής μου. Στην τροπολογία 3 έχουμε το κεντρικό και πιο επίμαχο θέμα και περιμένω να ακούσω τι γνώμη έχουν γι' αυτό οι συνάδελφοι. Η τροπολογία αυτή δίνει την δυνατότητα ο οργανισμός στο μέλλον να εισπράττει τέλη για κάποια από τα καθήκοντά του. Το δικαίωμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στο βασικό κανονισμό. Όμως ε, για πολύ περιορισμένα καθήκοντα τα οποία δεν... Ε, και η δυνατότητα αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Θα μπορούσα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μάλλον αυτό θα ήταν υπερβολικό αυτή τη στιγμή. Σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε ότι στα καθήκοντα του συμπεριλαμβάνεται και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των καθηκόντων των διαχειριστών δικτύων. Συμβάσεις για την παροχή ενέργειας που προσφέρονται στα χρηματιστήρια μπορεί να αποτελούν ε, αντικείμενο χειραγώγησης και σε σχέση με ακριβώς αυτό το τελευταίο θέμα. Είχα συζητήσει με τον Γενικό Διευθυντή του οργανισμού που μου είπε ότι θα πρέπει να εξετάζει ο οργανισμός κάθε μέρα συμβάσεις ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ την ημέρα. Και αν αυτό πρέπει να γίνει με σοβαρό τρόπο, αυτό θα είναι δύσκολο και γι' αυτό σημαντικό είναι να προβλέψουμε περισσότερο περιθώριο ε, στον οργανισμό να μπορεί να ε, χρεώνει τέλη και να έχει περισσότερο προσωπικό. Αυτή τη στιγμή ε, το, προσωπικό που έχει στη διάθεση του οργανισμού μου φαίνεται πολύ περιορισμένο για το καθήκον αυτό. 35 άτομα πλήρους απασχόλησης. Ε, υπάρχει οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίστοιχα καθήκοντα στον ε, τομέα τον χρηματοοικονομικό, ο οποίος ε, πράγματι χρεώνει τέλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, απλά θα εφαρμόσουμε αυτά που εφαρμόζει ήδη ο ΕΣΜΑ. Επίσης, ε, ο οργανισμός ε, θα πρέπει να ε, διατηρεί μητρό με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, TSO. Και υπάρχει εδώ ο φόβος οι επιχειρήσεις ε, να ζητήσουν καταχώρηση ε, στον ε, Acer προληπτικά, ακόμα και αν δεν είναι ακόμα κανονικοί διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς. Πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον Acer να χρεώνει τέλη. Γνωρίζετε ότι αυτό αυτό δεν είναι φορολόγηση, ε, προβλέπονται τα τέλη για την κάλυψη των ε, δαπανών του οργανισμού. Πιστεύω ότι αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο στη συγκεκριμένη περίπτωση και θα ανακουφίσει και σε κάποιο βαθμό τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη έχουμε το θέμα της ανεξαρτησίας ε, των ε, εποπτικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαγράψει μία φράση που της επιτρέπει τους εκπροσώπους της στο Συμβούλιο να τους δίνει οδηγίες. Αυτό δεν είναι Άρα πολύ ύποπτο, αλλά εάν το διαγράψουμε θα ισχύει το ίδιο που ισχύει και... Μάλλον εάν διαγράψουμε αυτή την φράση θα ισχύει και για, τους, ε, για τα άλλα μέλη του Συμβουλίου και γι' αυτό έχω επιλέξει εγώ διαφορετική διατύπωση. Προτείνω ο οργανισμός αυτός να έχει τη δυνατότητα που έχω προτείνει και κατά άλλες αναδιατυπώσεις για άλλους οργανισμούς. να μπορεί να ε, αναθέτει μεταφράσεις και σε άλλους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών, διότι το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης συχνά έχει υπερβολικό φόρτο ε, εργασίας, κάτι που οδηγεί σε καθυστερήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί ο οργανισμός να χρησιμοποιεί και άλλους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών. Επίσης προβλέπεται αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και, επίσης, και όλα αυτά σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης υπολογισμού βάση επιδόσεων. Ευχαριστώ πολύ. Merci pour ce rapport. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και για την έκθεση και τις τροπολογίες. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης, έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Σάρμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Γκάιερ για την επικοδομητική του προσφορά. Εγώ είμαι σκιώδης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και θα συμφωνήσω με την γραμμή την οποία ακολούθησε ο κύριος Γκάιερ για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας όπως επίσης και για την αιμονή του στην βασική αρχή του προϋπολογισμού του βασισμένου στα αποτελέσματα. Νομίζω όμως ότι οι ιδέες αυτές θα πρέπει να ε, προωθηθούν ακόμα περισσότερο και να ενισχυθούν και να ενσωματωθούν στα ίδια τα άρθρα του κανονισμού, στο άρθρο 32 και για τον προϋπολογισμό στο 33. Για το θέμα των τελών και της κάλυψης του κόστους των τελών, της χρηματοδότησης των τελών επίσης, εγώ είμαι δεκτικός σε κάποιες ιδέες, αλλά, αλλά και επιμένω σε αυτό, με την αίρεση ότι θα είμαστε σίγουροι ότι κάθε έσοδο το οποίο θα εισπράττει η υπερσία δεν θα δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με την, με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα της υπηρεσίας αυτής. Αυτά. Κατά τα άλλα υποστηρίζω την πρότασή σας. Ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο, δεν βλέπω κάποιον. Συνεπώς προσκαλώ τον εισηγητή μας ε, να κλείσει την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν διαφωνώ με τις προτάσεις του Πέτρη Σαβαρμά. Αν αυτό εξασφαλίζει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δεν έχω καμία αντίρρηση και κανένα πρόβλημα. Να δούμε πώς θα έχει διατύπωση των κειμένων που θα τεθούν προς ψήφιση. Και αυτά. Και χαίρομαι για την επικοδομητική συνεργασία που θα συνεχιστεί. Ωραία. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για τη γνωμοδότηση αυτή. 30 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι, το αργότερο. Η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή μας στις 30 Αυγούστου ενώ στην Επιτροπή Ήτρα που είναι αρμόδια επί της ουσίας στις 28 Νοεμβρίου θα ψηφίσουν. Ώρα ψηφοφορίας τώρα λοιπόν. Για να κάνουμε ένα τεστ, μια δοκιμή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Δεν έχω και την κάρτα μου. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Σας ευχαριστώ. Ας ψηφίσουμε λοιπόν τώρα πρώτη ψηφοφορία. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθμός 2 του Γενικού Προϋπολογισμού 2017. Για τροπολογία υπαριθμών 1 ψήφι υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 8 υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία υπερθμών 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 3 και 4 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτονται. Η τροπολογία βαθμό 5 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτονται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Η τροπολογία 7 είναι απαράδεκτη. Η τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές Η Τροπολογία βαθμό 9 υπέρ. Κατά. απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαρθμών 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επί του συνόλου του κειμένου ηλεκτρονικά παρακαλώ. Υπάρχει την ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ 2 κατά συγχαρητήρια ε, κύριε Σιγητά. Θα ξαναδώσω το λόγο στο Γιάννης Γκάιερ για τις μεταφορές πιστώσεων τμήμα 3. Δύο σχέδια μεταφορών. Πιστώσεων ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δώστε μου ένα λεπτάκι να βάλω μια τάξη στις σημειώσεις μου για να σας πω περί τίνος πρόκειται. Πρώτον, για να μην υπάρξει σύγχυση για την αρρύθμιση, η μεταφορά υπαριθμών 8 έχει να κάνει με αυτά που πρότεινε η κυρία Βάνα, την αίτηση για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και θα ε, ψηφιστεί πρώτο. Είναι λίγο περίεργη αρρύθμιση, δεν έχει γίνει κανένα λάθος. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω από τη μεταφορά πιστώσεων υπαριθμών 9. Θα ήθελα να σας τη συστήσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει παρουσιάσει με τρόπο αντιληπτό και κατανοητό τις οικονομίες που θέλει να κάνει, αλλά να πω εδώ ότι αυξάνεται το βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συντάξη των υπαλλήλων της και μέσω πρόθεσμα θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό, όχι αμέσως. Ε, ξέρω ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ασχολούνται με αυτό το θέμα και τους απασχολεί και τους ταλαιπωρεί. Στο επόμενο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να το ξαναδούμε. Κοιτάξτε, ο ρυθμός των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βγαίνουν στη σύνταξη αυξάνεται. Και επίσης αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής, πράγμα που είναι ε, θετικό και ο κόσμος ε, παραμένει συνταξιούχος περισσότερα χρόνια και καλά κάνει, αλλά είναι δύσκολη η χρηματοδότηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες, πολλά κράτη, καθώς γεράσει και ο πληθυσμός, αυξάνεται και η συνταξιοδοτική πίεση. Και στη Γερμανία ισχύει αυτό. Το γνωρίζουμε το πρόβλημα και θα πρέπει να δούμε, όχι βραβική πρόθεσμα, αλλά μέσω πρόθεσμα πώς θα αντιδράσει ο προϋπολογισμός. Μπορεί να υπάρχουν πιο ευθύς ε, λύσεις από το να λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Ακούσα και την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα ταμείο, ο αντίστοιχο του ταμείου για τους βουλευτές. Ε, τώρα δεν συμφωνώ ότι θα ήταν πιο ικανοποιητική λύση, γιατί στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού βλέπουμε ότι έχει λύματα το Ταμείο των Βουλευτών και δεν ξέρουμε πώς θα καλυφθούν. Δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση. Λοιπόν, ε, να ε, συμφωνήσουμε με τη μεταφορά πιστώσεων υπερθμών 9, με το 7, σε σχέση με θέματα που συζητήσαμε και το πρωί, αυτά που μας παρουσίασε η Ιντερκάντια Σάμπαλ, έχω πρόβλημα και το λέω έτσι πολιτικά αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει χρήματα από θέσεις του προπολογισμού στο τίτλο 4 εξωτερική πολιτική για να καλύψει απαραίτητες ε, πληρωμές για τη διευκόλυνση προς την Τουρκία και το θέμα του προσφυγικού. Ανάγκες που έχουν προκύψει από εκεί. Αυτό σίγουρα δεν είναι πρόβλημα, πλην όμως στα πλαίσια της κανονικής διαδικασίας του προϋπολογισμού, αρκετά συχνά έχουμε επικρίνει ότι το πρόβλημα είναι ότι ολόκληρος ο τίτλος 4 αποψηλώνεται για να πάνε αυτά τα λεφτά σε διάφορους σκοπούς, κυρίως στο διευκόλυνση με την Τουρκία. Εδώ έχουμε ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Η Ίντερ το είπε το πρωί. Υπάρχουν κάποια πράγματα όπου που μας ενδιαφέρει στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Προπολογισμού να υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση. Και αν βάζουν τόσο βαθιά το χέρι σε αυτές τις γραμμές του προπολογισμού για να τα δίνουν στη διευκόλυνση για την Τουρκία, θα πρέπει να μας τα εξηγήσει λίγο περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το έχει σκεφτεί και το έχει σχεδιάσει. Και θα παρακαλούσα να μην αποφασίσουμε σήμερα τη μεταφορά υπαριθμών 7, την 9, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο άλλο θα ήθελε το λόγο, η κυρία Γουάδια Ζάμπαλ. Θα είμαι σύντομη μετά τα σχόλια τα οποία έκανε ο κ. Γκέγερ για τη μεταφορά της έδρας. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη φάση εξετάζουμε διάφορες εκθέσεις τις οποίες διαπραγματευόμεθα το θέμα δεν είναι μόνο να προβλεφθεί μια αύξηση των όριων έτσι ώστε να φτάσουμε στα 35 εκατομμύρια μέχρι το 2020 εφόσον λέγεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποσά δεν ξέρω πως θα υπάρξει η μεταφορά αυτού του ποσού που είναι το διπλάσιο από αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να προβλέψουμε. Ε, Πρόκειται για ένα θέμα το, στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει πάρει μέρος στην συζήτηση. Το Συμβούλιο μόνο του προχώρησε στο μηχανισμό. Δεν ξέρω, αναζητεί βέβαια το Συμβούλιο να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες, αναζητώντας πιστώσεις δεξιά και αριστερά αλλά εμείς ε, σαν Επιτροπή Προϋπολογισμών αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τι χρήματα μπορούμε εμείς να προβλέψουμε για να εγκρίνουμε αργότερα αυτή τη μεταφορά. ο κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Σχετικά με την πρόταση του κύριου Γκάγερ θα συμφωνήσω μαζί του για τη μεταφορά υπαριθμε 9. Πρόκειται για μια πραγματικά ανάγκη θα έλεγα. Γύρω από το 7 τώρα θα ήθελα πριν ακούσω ξανά τον κύριο Γκάγερ να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πούνε το επίπεδο ανάγκης που έχουμε για αυτή τη μεταφορά. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξανανοίξουμε ένα μέτωπο με την Τουρκία για το θέμα των προσφύγων. Εάν υπάρχουν λοιπόν διαθέσιμα δημοσιονομικά μέσα, εγώ θα ήθελα να τα χρησιμοποιήσουμε. Πριν λοιπόν πάρω απόφαση για το 7, θα ήθελα να μου πούνε τον βαθμό ανάγκης και αναγκαιότητας γιατί δεν θα ήθελα η Τουρκία να αμφισβητήσει κάποια πράγματα από αυτά τα οποία αποφασίσαμε στα πλαίσια της δήλωσης. Βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε στην Ιταλία. Δεν θέλουμε δεύτερο μέτωπο, η κυρία Γκρέσλε. Μια ερώτηση έχω για τις συντάξεις. Βεβαίω να παίρνουν συντάξει οι υπάλληλοι, αλλά εδώ πρόκειται για αύξηση 3,3%. Και πού θα τα βρούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τοποθετηθεί. Δεν λέω να μην παίρνουν συντάξει οι άνθρωποι. Πρόεδρος, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Βλέπω ότι έχουμε 85 εκατομμύρια που πήραμε από τον προπολογισμό για την πολιτική ασφαλείας και προβληματίζομαι κατά πόσο είναι εύστοχο αυτό και ε, στο σχέδιο προπολογισμού που ψηφίζουμε είχαμε γράψει 300 εκατομμύρια και τώρα ερχόμαστε να βγάλουμε το 1 τρίτο, τα 85 εκατομμύρια. Γιατί την ανοίξαμε αυτή τη γραμμή. Έχω πραγματικά μείνει άναυδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας διαφωτίσει, παρακαλώ. Uh, thank you, Chair. Let, let me try. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, όσον αφορά την ερώτησή σας και την ερώτηση του κυρίου Ντεπρέ. Η μεταβίβαση των 85 ε, εκατομμυρίων, ε, η συνεισφορά δηλαδή του ΚΕΠΑ στην ε, χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία προβλεπόταν ήδη στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι την Άνοιξη. Δεν πρόκειται λοιπόν για νέο απρόβλεπτο στοιχείο. αποτελούσε τμήμα των 750 εκατομμυρίων που προβλεπόταν για τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες ε, στην Τουρκία το 2017. Και αυτά τα 85 εκατομμύρια, η συνεισφορά δηλαδή από τη γραμμή του προϋπολογισμού για ε, την ΚΕΠΑ, αποτελεί σημαντικό στοιχείο αυτής της δέσμης. Δεν είναι λοιπόν κάτι νέο. Προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι την Άνοιξη στο σχέδιο προϋπολογισμού και γι' αυτό υποθέτω κιόλα ότι εγκρίθηκε και τον Νοέμβριο. Η μεταφορά αυτή επίγει. Είναι επίγουσα η ανάγκη για αυτούς τους πόρους. Και έχω ήδη πείσει το Συμβούλιο όσον αφορά το ότι επήγει. Διότι, όπως θα γνωρίζετε, το Συμβούλιο αγαπά ιδιαίτερα αυτή τη γραμμή του προπολογισμού, Επήγει όμως, διότι αποτελεί μέρος ενό ενός χρηματοδοτικού πακέτου για σχολεία προκάτ για παιδιά προσφύγων στην Τουρκία, τα οποία θα πρέπει να είναι έτοιμα την 1η Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά. Επίσης θα χρηματοδοτηθεί νέο νοσοκομείο για σύρους πρόσφυγες. Η ανάγκη λοιπόν υπάρχει. Από την άλλη, αν ο κύριος Γκάιερ προτείνει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι την επόμενη συνεδρία, δηλαδή εντός του μήνα, δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει μεγάλη καταστροφή, διότι θα παραμείνετε εντός της προθεσμίας των έξι εβδομάδων όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε για τις ε, συντάξεις. Η αύξηση αυτών κατά 3,3% ακολουθεί και την αύξηση των ε, μισθών. Αυτή λοιπόν είναι η αιτήσια αναπροσαρμογή και για τους μισθούς ε, των υπαλλήλων και για τις συντάξεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γκρέσλε, ευχαριστώ πολύ. Στην αιτιολόγηση που μας έχετε δώσει λέτε ότι οι διορθωτικοί συντελεστές αυξάνονται αναπάντεχα. Πώς υπολογίζονται. Θα ήταν πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει και να μας δημοσιοποιήσει τον υπολογισμό. Μετά τη συνεδρίαση μπορείτε να μας εξηγήσετε. Πώς υπολογίζετε την άτα, την αύξηση των μισθών και των συντάξεων είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτοί οι συντελεστέ άλλαξαν σε τελευταία τροποποίηση του ε, κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας τα έχει στείλει, δεν ξέρω, ε, αμφιβάλλω ότι θα ενημερωθείτε. Κάθε χρόνο έχουμε εκπλήξει σε ό,τι αφορά τους δείκτες ε, αναπροσαρμογής των μισθών. Είναι ένα καλάθι που λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό στις διάφορες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μάλλον καλό για εκείνους που εργάζονται σε πρωτεύουσες όπου είναι σχεδόν μηδενικός ο πληθωρισμός, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα Μπορεί σε κάποιες χώρες να αυξηθεί σημαντικά η αμοιβή, αλλά ο κανόνας που έχει ε, αποφασιστεί μας ε, προκαλεί προβλήματα κάθε χρόνο. Όταν ε, εγκρίνουμε το σχέδιο προϋπολογισμού κάνουμε μια παραδοχή για ένα υπολογισμό και λίγους μήνες μετά ερχόμαστε και το αναθεωρούμε προς τα πάνω. Όλα αυτά τα μαζεύουμε στο λεγόμενο ραμασάζ στο τέλος, αλλά δεν είναι πολύ εύκολα ε, σε όρους δημοσιονομικούς. Και θα παρακαλούσα την κυρία Επίτροπο να λάβει ε, μέτρα. Το έχω ήδη ζητήσει, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Κύριε Γκρέσλε, κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη στα γαλλικά. Αυτά που μου λέτε τα ήξερα. Εγώ θέλω τον πραγματικό υπολογισμό. Ε, το, το συγκεκριμένο, πώς υπολογίζεται στην πράξη κάθε χρόνο αυτή η αναπροσαρμογή και γιατί; 1η Ιουλίου του 2016 συγκεκριμένα γιατί θα ήθελα να συγκρίνω τη νέα μέθοδο με την παλαιά η οποία άλλαξε το 2014. Γι' αυτό έχει σημασία. Γιατί εδώ δεν έχουμε διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα θα σας ε, κοινοποιηθεί το συντομότερο αυτή η πληροφορία. Κύριε Γκάιερ έχετε να προσθέσετε τίποτα. Ε, να ψηφίσουμε. Ωραία, ψηφίζουμε. Τη μεταφορά υπαριθμών 7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πρόβλημα να αναβληθεί, μας είπε η ψηφοφορία. Μπορώ να θεωρήσω ότι συμφωνείτε με τον εισηγητή. Να αναβληθεί η ψηφοφορία της μεταφοράς υπαριθμών 7. Ωραία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την μεταφορά υπαριθμών 9. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Όχι από ό,τι βλέπω. Λείπουν ακόμα μερικοί. Vous Πέρασε, αφού δεν θέλει να ψηφίσει. Εγκρίνεται μεταφορά 17 ψήφοι υπέρ και μία ψήφος κατά. Λοιπά τμήματα. Κύριε Τάραντ. Τρεις μεταφορές έχουμε εδώ που μπορεί και να μην ψηφιστούν. Αν δεν διαφωνεί κανείς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Τάραντ. Ε, thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη από την ε, Επιτροπή, διότι θα δαπανίσουμε χρόνο σε κάπως ασήμαντα ποσά. Έχουμε λοιπόν τρεις ενημερώσεις από την Επιτροπή των Περιφερειών που συμπεριλαμβάνονται στα 162.000 τα πρώτα 110.000 για το πρώτο, 10 ε, για ε, την δεύτερη και 32 για την τρίτη. Ενώ η ΕΟΚΕ δαπανεί περίπου 225 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν είναι λοιπόν πολύ χιλιάδες το χρόνο. Δεν είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Δείχνει όμως πώς λειτουργούν αυτά τα θεσμικά όργανα. Και θα ήθελα να σχολιάσω την πρώτη μεταφορά. Προβλέπεται μεταφορά από τη γραμμή 264, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό. Αν λάβουμε υπόψη τον στόχο της μεταφοράς αυτής. Ε, οι πιστώσεις ήταν σχεδόν 19.000 για το 2017, κάτι που ήταν ε, σχεδόν 25% λιγότερο από ό,τι είχε ζητηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέκοψε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού, κάτι το οποίο τελικά συμφωνήθηκε. Κατά τη γνώμη μου, όταν γίνεται περικοπή της γραμμής του προϋπολογισμού, τότε θα πρέπει το θεσμικό όργανο να προσαρμοστεί στις νέες πιστώσεις και να αναπρογραμματίσει τις δραστηριότητές του. Η Επιτροπή των Περιφερειών όμως αποφάσισε να συνεχίσει να προχωρήσει στις προγραμματισμένες ε, δράσεις και να ε, υποβάλει αίτηση για επιπλέον 148.000. Κάτι που δείχνει σαφή έλλειψη προληπτικής εποπτείας εφόσον ε, ο υπάρχον προϋπολογισμός εξαρτηθεί ήδη στα μέσα της χρονιάς. Γι' αυτό διστάζω όσον αφορά την ε, σύσταση αυτή. 13 σελίδες εξηγήσεων μου έστειλαν και είναι αρκετά ασαφής. Ε, δεν γνωρίζω πολύ καλά η, η Επιτροπή των Περιφερειών πώς συμμετέχει σε διάλογο με τους Ευρωπαίους πολίτες για να δώσει ε, στοιχεία σχετικά με νομοθετήματα. Επίσης, η διάσκεψη των Προέδρων ε, επισκέφτηκε η Ιταλική περιφέρεια που είχε πληγεί από σεισμό. Καταλαβαίνω ότι οι σεισμοί δεν προγραμματίζονται, αλλά αποτελεί ηρωνία δεδομένου το πόσο ε, θα, μπορούσε, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους πληγέντες. Και επίσης ε, θέλουμε να αποφύγουμε τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα ε, που έχουν οδηγήσει στο Brexit ε, και που συζητώνται γενικά και για άλλες χώρες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξουμε πολύ πώς πανούμε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη ενημέρωση συνδέεται με την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πληρωμές ε, για βρεφοκομεία. Και και σταθμού. σταθμούς. Αναφέρεται η αύξηση του διαλόγου με τους πολίτες ε, και η εντατικοποίηση δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Ναι, καταλαβαίνω τι προσπαθούν να πούν, αλλά Θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών. Και τέλος, ...32.143 ευρώ προβλέπονται για ε, συμπληρωματικές υπηρεσίες ε, για τη μετάφραση και καλύπτουν εξωτερικές ανάγκες μετάφρασης. Ενώ η γραμμή του προϋπολογισμού μιλάει για εξωτερική βοήθεια ή ε, συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής ε, της Επιτροπής των Περιφερειών, ε, καθώς και χρηματοδότηση ενός νέου συστήματος διαχείρισης της μετάφρασης. Και πάλι θυμάμαι ότι είχαμε πολύ δύσκολες συζητήσεις σχετικά με την συγκέντρωση των υπηρεσιών μετάφρασης και άλλων υπηρεσιών και καταλήξαμε σε μια πολύ συγκεκριμένη λύση για την Επιτροπή των Περιφερειών που μάλλον δεν ταιριάζει με το σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να συνοψίσω λοιπόν, πιστεύω ότι το σύστημα των μεταφορών και το γεγονός ότι η Επιτροπή των Περιφερειών ε, συνεργάζεται με την ΕΟΚΕ Αυτά τα εκμεταλλεύεται η Επιτροπή των Περιφερειών με τρόπο που δείχνει ότι πιθανότατα τα δύο αυτά θεσμικά όργανα να έχουν προβλήματα όσον αφορά την εποπτεία. Και γι' αυτό ως εισηγητής για τα άλλα τμήματα για το 2017... Συμμερίζομαι και τις θέσεις ε, του εισηγητή και συνεισηγητή. Πιστεύω ότι ίσω να, έχουν, ίσως να είναι εκείνοι πιο τυχεροί όσον αφορά την επιλύση των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Αυτό τι σημαίνει κύριε Σιγητά, θέλετε να αναβληθεί η απόφαση περιμένοντας συμπληρωματικές πληροφορίες. Μάλιστα, ακριβώ αυτό. Προηγουμένως όμως θα δώσω το λόγο στη Μόνικα Χόλμαγια. Κύριε Πρόεδρε, συζήτησα με την Επιτροπή Περιφερειών και για την κτηριακή πολιτική και άλλα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Παρακαλώ να δείξουμε λίγη κατανόηση. Δεν έχουν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό και όταν γίνονται κάποιες μετατοπίσεις και αλλαγές. Τις βρίσκουμε πολύ γρήγορα μπροστά μας στην Επιτροπή εδώ προϋπολογισμών ακριβώς επειδή είναι μικρός ο προπολογισμό τους. Προσοχή θα πούμε εμεί στον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών που θα ταξιδεύσει και που δεν θα ταξιδεύσει. Το ίδιο ισχύει ε, ε, και για τους ευρωβουλευτές. Δηλαδή, αν πάμε εμείς σε μια περιοχή, δεν τη βοηθάμε ιδιαίτερα. Ε, δεν αλλάζει η κατάστασή τους, η σεισμόπληκτη. Προφανώς δεν έχουμε μεγάλο όφελος από την παρουσία μας εκεί, αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντικό να ταξιδεύουμε και να πηγαίνουμε στις διάφορες περιφέρειες. Ας πούμε, από τη δική μου περιφέρεια ε, πηγαίνει το ΤΕΧΑΒΕ που είναι η τεχνική βοήθεια σωστικά συνεργεία από τη Γερμανία στις σεισμόπληκτες περιοχές και δεν επιβαρύνεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αλλά χρησιμοποιούνται οι διάφορες υποδομές επιτόπου. Αν θέλετε μπορούμε να σε ενημερώσουμε περαιτέρω. Μπορεί κανεί να είναι υπέρ ή κατά τη επιτροπή των Περιφερειών, αλλά τα επιχειρήματα ειλικρινά ισχύουν και για εμά. Δηλαδή αν θα μεταβεί η διάσκεψη των Προέδρων των Περιφερειών, ισχύει και για του Ευρωβουλευτέ αυτό. Μάλιστα, δεν θέλει. Έχουν ζητήσει άλλοι το λόγο. Κύριο Σάβαμα, να προσθέσω σύντομα ότι προσωπικά το θέμα δεν είναι η Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι θέμα αρχή. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρά ποσά, είναι αλήθεια. Από την άλλη όμως θα μπορούσε να πει κανείς ότι έφτασε η στιγμή να στέλνουμε τα σωστά μηνύματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εμένουμε σε αυτή την λογική ακόμα περισσότερο όταν υπάρχουν έστω κάποιες αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα πράγματα, θα πρέπει να στέλνουμε τα μηνύματα και να παίρνουμε όλες τις πιθανές εξηγήσει και τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε, έτσι ώστε τον επόμενο χρόνο να μην συμβούν ξανά τέτοιου είδους συμβάντα. Νομίζω λοιπόν ότι έχει δίκιο η συγητής. Nous avons parmi Έχουμε δύο εκπροσώπους της Επιτροπής των Φεριών, τον κύριο Πέντευσεν και τον κύριο Κρόνμπερξ. Τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών θα ήθελαν να, εκφραστούν ε, σε σχέση με τις ερωτήσεις του κυρίου Τάραντ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πρώτες τρεις μεταφορές είναι μεταφορές οι οποίες έχουν σαν στόχο την στήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έχουν καθοριστεί, έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν σαν παράδειγμα και κάποιες εκπεφασμένες επιθυμίες και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως επίσης ε, και ε, να λάβουμε υπόψη μας, λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά τα οποία έχει ζητήσει ο κύριος Τάσκ. Το θέμα δεν είναι να προβλέπει κανείς απόλυτα τα πράγματα, γιατί πολλές φορές οι πολιτικές συνθήκες αλλάζουν και με μεγάλη ταχύτητα και εμείς είμαστε αρκετά ευέλικτοι προσπαθώντας να δείξουμε ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτά τα οποία θέλει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτά όμως δεν καθορίζονται δύο χρόνια νωρίτερα. Αν πούμε πριν δύο χρόνια ότι θα κάνουμε μετά από δύο χρόνια κάτι, ε, μπορεί να μεσολαβήσει κάτι και δεν θα μπορούμε να το καλύψουμε. Τώρα, σχετικά με την 264, γραμμή 264. Αυτή είναι μια απόφαση που ελήφθη μετά από τη συμφωνή των πολιτικών ομάδων και είναι κάτι το οποίο ζητήθηκε και από τον πρόεδρο Τάσκ. Διευκολύνει την επικοινωνία στο εσωτερικό της πολιτικής οικογένειας, αν θέλετε. Είναι κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε επίσης και από τον ίδιο τον κύριο Ταγιάννη. Εμείς έχουμε ήδη ξεπεράσει τα ποσά που είχαμε στη διάθεσή μας για το 2017 και οι δαπάνες αυτές υπάρχουν γιατί χρειάζεται να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο οι συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και όχι να μειωθούν. Τώρα για, το... για μια στιγμή. Να πω ότι οι υπηρεσίες έχουν επιβεβαιώσει ότι θα χρειαστούν περισσότερες πιστώσεις στο 162 αν θέλουν να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες σε διάφορους τομείς όπως ε, συναντήσεις διαφόρων ομάδων εργασίας και διαφόρων οργάνων της Επιτροπής Περιφερειών που είναι υποχρεωτικές λόγω ανηρημένων υποχρεώσεων αλλά δεν ασχολούνται, δεν καλύπτουν αν θέλετε τις κεντρικές δομές της Επιτροπής. Τώρα για το Reflecting Europe ο πρόεδρος Τάσκ έχει ζητήσει από, το, από την Επιτροπή να εμπλακεί σε βαθύτερο διάλογο με τους Ευρωπαίους πολίτες έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς λοιπόν για να διευκολύνουμε αυτό τον διάλογο στις περιφέρειες απαιτείται λογιστική ε, βοήθεια και για την επικοινωνία και για το γραφείο του Προέδρου και είναι κάτι που έχει υπογραμμιστεί από, τις, ε, από όλα τα θεσμικά όργανα και τους γενικούς διευθυντές Ο Διευθυντής λοιπόν για την επικοινωνία έχει στον τομέα της εξωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης εντατικοποιήσει την δράση της γενικής του ε, διεύθυνσης. Και μάλιστα στα πλαίσια της απαλλαγής για το 2016 ε, έχει η δράση του ειδωθεί με ε, πολύ θετικό τρόπο και η συνέχιση της δράσης αυτής θεωρείται ότι είναι ζωτική. Λόγω ακριβώς της βεβαρημένης πολιτικής ατζέντα και της ισχυρής κινητοποίησης των θετικών οργάνων έτσι ώστε να προωθήσουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προς τις εκλογές του 2019 και στα πλαίσια των συζητήσεων για το νέο ε, πολιετές δημοσιονομικό προβλέπεται για το 17 και 18 μια σωστή συνοδεία της πολιτικής διαδικασίας έτσι ώστε η Ευρώπη να έρθει πιο κοντά στους πολίτες και να υπογραμμιστεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό σημαίνει νέες δημοσιονομικές ε, διαθεσιμότητες και νέες συναντήσεις οι οποίες προϋποθέτουν και τη συμμετοχή του προσωπικού. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να τα σχεδιάσουμε όλα εκ των προτέρων. Θα ήθελα να πω να σας ζητήσω να λάβετε υπόψη ότι η μεταφραστική υπηρεσία είναι κάτι το οποίο μοιραζόμαστε με την οικονομική και κοινωνική. Και η Επιτροπή σας έχει ήδη εγκρίνει ε, ε, κάποιες επιπλέον δαπάνες για το ΕΚΟΣΟΚ. Μέχρι τώρα δηλαδή έχετε κάνει τη μισή δουλειά και γι' αυτό σας ζητάμε να μας ε, επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, ο κύριος ε, Γκάιερ. Ε, συγγνώμη, ο κύριος Τάραντ. Εμένετε στο αίτημα σας για αναβολή. Σε ό,τι αφορά το τρίτο, είναι γεγονός ότι εγκρίναμε ε, το αίτημα ε, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και αυτή είναι η δεύτερη ε, δόση. Δεν έχω αντίρρηση να το εγκρίνουμε, αλλά τι θα πει meaningful political communication. 50.000 ευρώ δηλαδή για να έχουμε ουσιαστική πολιτική επικοινωνία. Και ποιος το ορίζει αυτό και ποιος το επαληθεύει. Ο εσωτερικός ελεγκτής που μπορεί να ταξιδεύσει εκεί πληρώνοντας 500 ευρώ και τα γραφεία τύπου. Εγώ βλέπω τι κάνει η Επιτροπή. Στέλνουν κόσμο για να κάνει αναρτήσεις στο Twitter ή στο Facebook. Αυτό είναι η πιο ουσιαστική πολιτική επικοινωνία προς τους πολίτες. Ας τους καλέσουμε εδώ τους πολίτες αυτό θα έχει μεγαλύτερο νόημα. Γι' αυτό χρειάζομαι περισσότερη ενημέρωση. Δεν είναι απλώ μια πολιτική επιταγή. Εντάξει, άρα ζητάτε αναβολή. Ναι, για τις δύο πρώτες μεταφορές χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, λέει ο συγητής. Ωραία. Ρωτώ την Επιτροπή μας. Συμφωνείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, να αναβληθεί η απόφαση για τις δύο αυτές μεταφορές. Υπέρ της αναβολής. κατά αποχές βάλετε λοιπόν. κυρία Χολμάια. Le report vous... Α, η αναβολή λοιπόν ισχύει. Και για τις τρεις ε, ε ψηφίσαμε τώρα. Όχι. Είχαμε τρεις μεταφορές. Η NF1, η NF2 το 2017 και η NF3. Θεωρώ ότι ισχύει και για τις τρεις μεταφορές πιστώσεων η ψηφοφορία. Α, επανάληψης. Λοιπόν, για την πρώτη. Ε, Δράσεις των πολιτικών ομάδων, ποιος είναι υπέρ της αναβολής της πρώτης μεταφοράς. Μα και για τις τρεις δεν ψηφίσαμε. Νόμιζα ότι ψηφίσαμε για τις τρεις. Όχι, για τις δύο. Καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, ψηφίσαμε και τα τρία, πάει και τελείωσε. Είμαστε εντάξει. Κυρία Χόλμαια, από κτίρια, πώς πάμε. Έχουμε αιτήσει ε, μεταφοράς πιστώσεων για τις κτηριακές υποδομές. Κοιτάξτε, στην Κολομβία λέει είναι ένα κτίριο, ε, το οποίο ε, μόλις μας έφτασε ως αίτηση, θέλει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία να αγοράσει και τον πέμπτο όροφο σε ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιεί ήδη και ενδρεύει. Ε, θα το κοιτάξω λίγο γιατί η Κολομβία δεν είναι και ασφαλέστερη χώρα ε, γιατί δεν έχουμε και μεγάλη πληροφόρηση ή προειδοποίηση, τίποτα. Πρώτη φορά το βλέπω, θέλω να το μελετήσω παρακαλώ και την επόμενη φορά μπορώ να μιλήσω και γαλλικά αν θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. Alles gut, Όλα καλά, να τα ξαναπώ από την αρχή. Λοιπόν, έλεγα ότι για την Κολομβία θέλω να το κοιτάξω λίγο και να σας πω την επόμενη φορά περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Και έχω την εξής παράκληση, αγαπητέ Πρόεδρε. Να γράψουμε στην ημερήσια διάταξη και το κτίριο Polaris Park. Δυόμιση-τρία χρόνια το παρακολουθώ και λυπάμαι πάρα πολύ που αναβάλλεται συνεχώς χωρίς να ενημερώνεται η Επιτροπή Προπολογισμού για τη μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική του Κοινοβουλίου για τα κτίρια στις Βρυξέλλες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε σε μεγαλύτερο βάθος με το θέμα αυτό, γιατί ένα τμήμα του κτηρίου θα πρέπει επιγόντως είτε να εξηγιαθεί, είτε να ανακαινιστεί, είτε να ξαναχτιστεί, ξέρω εγώ, θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να μας ενημερώσει το Προεδρείο. Τι γίνεται εκεί στι στις για να μην εξαρτώμαστε από τα δημοσιεύματα του τύπου που είναι τα μισά ε, ακριβή και τα άλλα μισά ανακριβή. Και τίθεται και θέματα ασφάλειας, ε, να δούμε τι γίνεται με τις μελέτες και τις γνωμοδοτήσεις που ίσως δεν θα πρέπει να συζητούμε δημόσια, αλλά να μην μαθαίνουμε τα πράγματα από τις εφημερίδες, αλλά στην Επιτροπή μας ε, κανονικά και επίσημα να ενημερωνόμαστε για την επόμενη πρόοδο. Γιατί πάνε τρία χρόνια που δεν μας ενημερώνουν και μπλοκάρουν διάφορα πράγματα, για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω και θα παρακαλούσα να εγγραφεί στη μερική διάταξη. Και κλεισμένο το θηρόν, λέω. Et Πολύ ωραία. Επ' ευκαιρία, καλό θα ήταν να γνωρίσουμε και πόσο θα στοιχήσει η ανακαίνιση αυτού του μουσείου που αγόρασε το κοινοβούλιο για συμβολικά ένα ευρώ, αλλά δύο-τρία εκατομμύρια στήχησε η ανακαίνισή του. Ε, αυτά θα πρέπει να τα μαθαίνει η Επιτροπή Προπολογισμού για να γνωμοδοτεί κιόλα. Παρακάλεσα και στο παρελθόν να μας ενημερώνει κάθε φορά το κοινοβούλιο ότι ό,τι αγοράζουμε συμβολικά προς ένα ευρώ να ξέρουμε τι μελλοντικό κόστος θα έχει αυτό και ισχύει και για τα τρία θεσμικά όργανα. Εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί καθόλου σωστά. Κανονικά θα έπρεπε το Προεδρείο να τα κάνει αυτά. Très euh, il a pas de Θαυμάσια. Άρα δεν έχουμε εδώ να πάρουμε απόφαση. Θα κάνουμε ένα μικρό δίλεπτο τεχνικό διάλειμμα γιατί η επόμενη ενότητα είναι και κλεισμένα των θυρών. Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή να αποχωρήσουν. Διακοπή